Ε, ήταν μια πολύ επιτυχής πρωτοβουλία των πολιτών και ο πρόεδρος των Σοσιαδημοκρατών είχε αποστείλει και Διακόπτει ο Πρόεδρος. Με συγχωρείτε να σας διακόψω. Παρακαλώ πρώτα να καλύψουμε τα διοικητικά πρώτα και μετά θα λάβετε τον λόγο για αυτό το θέμα το οποίο ζητήσατε. Κυρίε και κύριοι, έχουμε αρκετά διοικητικά θέματα που πρέπει να τα καλύψουμε, να τα διευθετήσουμε και μετά θα περάσουμε στα διαδικαστικά. Τετάρτη 2 Απριλίου είχαμε και μία σύσταση για την Επιτροπή Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων για μία απόφαση <clears throat> να μην υπάρξουν κάποιε ενστάσεις ε, για τον κανονισμό όσον αφορά τη συμπλήρωση του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους, ε, τα πιο ευάλωτα άτομα. Για αυτή τη σύσταση δεν υπήρξαν ενστάσεις και θεωρείται ότι εγκρίνεται. Αύριο λοιπόν στο εγκεκριμένο κείμενο θα δημοσιευθεί ω έχει. Σύμφωνα με το άρθρο 216 του κανονισμού μας θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι για τα διορθωτικά <clears throat> που ε, για την ε, Δευτέρα Απριλίου είχαν δοθεί δεν υπήρξαν κάποια άλλα διορθωτικά και έτσι θεωρούνται αυτά ότι εγκρίνονται τα διορθωτικά αυτά οι αρμόδιες ε, επιτροπές έχουν διαβιβάσει διορθωτικά σε τέσσερα κείμενα. Όσον αφορά το άρθρο 218 εδάφιο 4, θεωρείται ότι αυτές οι διορθώσεις εγκρίνονται ή θεωρούνται έγκυρες αν μέσα σε 24 ε, ώρες από μια κοινοβουλευτική ομάδα ή τουλάχιστον 40 μέλη δεν έχουν υπάρξει κάποιες ενστάσεις ε, και έτσι λοιπόν θα βρείτε αυτά τα κείμενα στα πρακτικά αυτής της συνεδρίασής μας. Σύμφωνα με το άρθρο 216 εδάφιο 3, η Επιτροπή, 211 ε, εδάφιο 3, η Επιτροπή η Συνταγματικών Υποθέσεων προβλέπει τα εξή. Το άρθρο 166, άρθρο 167, παράγραφος 1 και το άρθρο 195 εδάφιο 3 για την ονομαστική ψηφοφορία και για το άρθρο 6β εδάφια 2 και το 7 παραγραφή 3, 6 και 8